Κλείνοντας θα ευχαριστήσω και τους τρεις εισηγητές ε, και ελπίζω ότι θα επηρεαστούν ε, οι ε, διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Σας ευχαριστούμε κύριε Κάζακ. Από πλευράς των Πρασίνων, ο συνάδελφος Τέιλορ.